Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ε, ζητώ συγγνώμη και για τη δική μου καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε καν απαρτία, αλλά έχουμε την ε, συνεδρίαση για την προετοιμασία της επόμενης ΚΟΖΑΚ, επομένως είναι αιτιολογημένοι όσοι λείπουν. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η συνεδρίαση μαγνητοσκοπείται και μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Πρώτο σημείο λοιπόν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχω να σας ε, επισημαίνω αρκετές αλλαγές. Καταρχάς, σήμερα θα πρέπει να ψηφίσουμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων θα λάβει υπόψη τη γνωμοδότησή μας ε, αύριο ε, στη δική της ψηφοφορία. Έχουμε πρόβλημα όμως για τα δημογραφικά στατιστικά, γιατί δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε συμβιβασμό. Θα ακούσουμε και την άποψή σας, αλλά λογικά θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία για αύριο το πρωί στις 10, εάν είμαστε όλοι στην ώρα μας, αφού θα έχουμε ακούσει και την άποψη των συντονιστών. Οι συντονιστές δεν μπορούν να συνεδριάσουν σήμερα όπως είχε προβλεφθεί διότι απουσιάζει και ο κύριος Γκουαλτιέρη και ο κύριος ε, ε Τρασκόφσκι. Ο κύριος Γκουαλτιέρη νομίζω ότι είναι στο Δουβλίνο, ο κύριος Τρασκόφσκι δεν ξέρω ακριβώ που είναι. Έχει πάντως και αυτός κάποια προβλήματα και επομένως επειδή απουσιάζουν δύο συντονιστές και μάλιστα ε, του δικού τους ε, κύρους. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνεδρίαση των συντονιστών. Θα κάνουμε λοιπόν αύριο 9 με 10 συνεδρίαση των συντονιστών και στις 10 ακριβώ, αν δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις από πλευρά συντονιστών, μπορούμε να ψηφίσουμε το θέμα των δημογραφικών στατιστικών και κατόπιν μπορούμε να περάσουμε στο σύνηθες ε, πρόγραμμά μας και να ακούσουμε γύρω στις 11 και την Ιρλανδή Υπουργό. Αν συμφωνείτε λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τώρα την έκθεση Γιαννάκου για τα πολιτικά, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, επειδή οι τροπολογίε είναι διαθέσιμε μόνο στην ε, αρχική γλώσσα, καλό θα ήταν να κάνουμε τώρα μια αρχική ανταλλαγή απόψεων και γενικέ παρατηρήσει τη εισηγήτρια και να διευκρινίσουν και τι τροπολογίε όσοι τι κατέθεσαν εν ώψη και πιθανών διαπραγματεύσεων για συμβιβαστικέ τροπολογίε. Νομίζω ότι σας τα είπα όλα. για το σχεδιο εξεση έξεσης ε, Τραφσκόφσκι-Γουαλτιέρη για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου, αλλά και γι' αυτό η, την έκθεση δεν είναι ακόμα διαθέσιμε όλες οι μεταφράσεις. Υπάρχει όμως περίπτωση μέχρι αύριο να έχουμε κάποια κείμενα μεταφρασμένα. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν παρατηρήσεις, θέλετε να πείτε κάτι κύριε Γκερέρο, παρακαλώ. Ναι, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά γιατί είναι και η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για το 2013. Η πολιτική ομάδα συμφωνεί πολύ με τα όσα μας προτείνεται, δηλαδή να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τις δημογραφικές στατιστικές για αύριο το πρωί και να αποφασίσετε κατά πόσον υπάρχει συμφωνία στη συνεδρίαση των συντονιστών που θα γίνει πριν ε, ξεκινήσουν οι εργασίες της Επιτροπής. Συμφωνώ λοιπόν για την αναβολή για αύριο το πρωί και να αφήσουμε την απόφαση στα σχέδια των συντονιστών οι οποίοι θα συνεδριάσουν αύριο το πρωί να ψηφίσουμε στη συνέχεια και την έκθεση του κυρίου Ράνχελ για λόγους χρονοδιαγράμματος και να κάνουμε και ανταλλαγή απόψεων και εξήγηση των τροπολογιών για την έκθεση Γιαννάκου. Ουσιαστικά λοιπόν στηρίζω την πρότασή σας κύριε Πρόεδρε. κύριος Yes, ε, Ναι. Καλησπέρα σας. Νομίζω πως δεν έχουμε άλλη επιλογή Εκτό από το να αλλάξουμε τη μέρη σχεδία αλλά το θέμα είναι πως θα έχουμε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε το περίπλοκο ζήτημα της κατανομής των εδρών. Και δεν είναι σωστό να στριμώξουμε αυτή τη συζήτηση σε μισή ώρα. Κάπου τόσο, εν πάση και αν είναι αναγκαίο λόγω της ε, σημασίας ε, του να λάβει το Κοινοβούλιο άμεση απόφαση νομίζω πως θα καταλήξουμε σε μια κατεπίγουσα συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Οι συντονιστέ λοιπόν αύριο το πρωί θα μπορέσουν να συζητήσουν και αυτό το ζήτημα και να δούμε αν ε, θα πρέπει να γίνει και μια έκτακτη συνεδρία επί του ζητήματο. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν άλλε παρατηρήσει για το σημείο αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο υπαρχόν 3, έγκριση των πρακτικών τη προηγούμενη συνεδρίαση. Έχουμε τα πρακτικά τη συνεδρίασης της 19 η Νοεμβρίου του 2012 και είναι διαθέσιμα και ως συνήθως αν δεν υπάρχουν ενστάσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο σημείο 4 Ευρωπαϊκές Δημογραφικές Στατιστικές. Εγώ είμαι συντακτής της γνωμοδότησης και όπως σας είπα δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει στε συμβιβασμό. να δούμε αν μέχρι αύριο το πρωί καταφέρουμε να έχουμε μια συμφωνία. Ιδάλλως θα πρέπει ή να ψηφίσουμε ή να αναβάλουμε τη συζήτηση. Θα το δούμε αύριο το πρωί. Όποιο θέλει τον λόγο για το θέμα αυτό, για να συζητήσουμε ίσως και λίγο καλύτερα τις τροπολογίες, μπορεί να λάβει το λόγο. Νομίζω ότι είναι και εδώ και ο κύριος Εντουάρδο Βαρέρο Καπελό, ο οποίο είναι διευθυντή ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αρμόδιου τμήματο και θέλει να ε, εκφράσει την άποψή του για το θέμα αυτό. Θέλετε να λάβετε πρώτα το λόγο εσεί, λοιπόν, ή να δώσουμε πρώτα το λόγο στου βουλευτέ, όπω ε, γίνεται συνήθω. Ο κύριο Γκερέρο, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι για το θέμα επί της ουσίας, δηλαδή να βρεθεί μια συμφωνία για όλα όσα εξακολουθούν να μας χωρίζουν. Ουσιαστικά πρόκειται για την τροποποίηση του άρθρου 4. Αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο εργασίας αύριο από τους συντονιστές, ονόματος των πολιτικών ομάδων. Όμως θα ήθελα να εκφράσω μια ανησυχία που έχουμε από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών γιατί εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για μια συμβιβαστική τροπολογία στην οποία αρχικά δεν θεωρείται ότι θα είχε έμπαινε η αναφορά στον αντίκτυπο στην ειδική πλειοψηφία εντός του Συμβουλίου. Όμως, λάβαμε κάποιες πληροφορίες ότι για νομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν ή δεν ε, πρέπει να αποκλείσουμε αυτή την αναφορά και επίσης ε, μια τέτοια αναφορά θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να εμποδίσει προσωρινές μεταναστεύσεις που γίνονται από υπηκόους κάποιων χωρών να έχουν αντίκτυπο στο δικαίωμα ψήφου, στην ποσόστοση ψήφου των αντίστοιχων χωρών. Ανακοινώνω λοιπόν ότι ένα τμήμα της δουλειά που θα πρέπει να γίνει για να προχωρήσουμε αύριο στην ψηφοφορία θα ήταν πώς να διατηρήσουμε αυτή την αναφορά στην ειδική πλειοψηφία, στη ψηφοφορία του Συμβουλίου και ταυτόχρονα να εργαστούμε επί της συμβιβαστικής τροπολογίας που, επί της οποίας είχαμε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ίσως λοιπόν γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο οι γραμματείες των πολιτικών ομάδων μπορούν να κάνουν ε, αυτή τη δουλειά πριν από τη συνεδρίαση των συντονιστών αύριο το πρωί, απόψε δηλαδή. Ο κύριος Ντάφ. Κύριε Πρόεδρε, οι φίλοι είναι υπέρ ε, της πρότασης της ε, Κομισιόν ουσιαστικά. Δεν βλέπουμε κάποιο λόγο για να περιπλέξουμε ένα ζήτημα τεχνικό. Και σε ένα πνεύμα συμβιβασμού, έτσι ελπίζω να το έχετε κατά αυτό. Um, Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τις διάφορες εξυπνάδες ε, περιστατιστικής γιατί τα έχουμε ξανακούσει αλλά όσες φορές ε, και αν τις έχουμε ξανακούσει έχουν και κάποια αλήθεια. Η στατιστική από τη φύση της περιλαμβάνει την κατασκευή κατηγοριών που μπορεί να συγκριθούν με άλλες κατηγορίες που έχουν κατασκευαστεί χωριστά και μετά μπορούμε να δούμε τυχόν συσχετισμούς. Όταν έχουν συλλεγεί λοιπόν προσεκτικά τα ατιστικά στοιχεία ε, μπορούν να θεωρηθούν ε, αντικειμενικά και μάλιστα στο επεξηγηματικό σημείωμα εδώ πέρα λέει πως πρέπει να συμμορφώνται σε κάποιες προδιαγραφές αμεροληψίας. Αλλά βεβαίως οι κατηγορίες των δεδομένων είναι υποκειμενικές και κατά κάποιον τρόπο προϋποθέτουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν δείτε τις τροπολογίες ε, που έχουν προταθεί υπάρχουν αρκετά τέτοια παραδείγματα και σε πολλές περιπτώσεις οι κατηγορίες θα επιλεγούν έχοντας κατά νου ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα το επεξηγηματικό σημείο μας σε ένα άλλο σημείο κάνει λόγο για την ανάγκη ποιοτικών στατιστικών στοιχείων για να σχηματιστούν επιχειρησιακοί στόχοι. Με άλλα λόγια, έχουν υπόψη κατά νου δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα πριν επιλεγούν οι κατηγορίες. Οπότε τα στατιστικά στοιχεία είναι σαν μια αντικειμενική απάντηση σε μια υποκειμενική ερώτηση. Και άρα δεν έχουν και ιδιαίτερη αξία από αυτή την έννοια δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν το λόγο. Έτσι λοιπόν θα παρακαλέσω τον κύριο Μπαρέδο Καπελό να πάρει το λόγο για να μας πει ποια είναι η θέση της Κομισιόν για το ζήτημα αυτό των στατιστικών δημογραφίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρέδο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα και τον αντικαθιστώ από την κύριο Στάτα. δεν αμφισβητείται η ανάγκη να έχουμε στατιστικές για δημογραφική για δημογραφικούς λόγους, έτσι λοιπόν, ε, ε, χρησιμεύουν για την ειδική πλειοψηφία, για τη διαφορετικά ταμεία, για να δούμε τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών ή, για παράδειγμα, για τη στρατηγική αηφόρου ανάπτυξης. Υπάρχει ανάγκη για αυτόν τον κανονισμό, γιατί αυτά τα δεδομένα συλλέγονταν βάσει συμφωνία κυρίων εδώ και πολύ καιρό. Έτσι λοιπόν, κάθε χρονό Eurostat ήδη διαβιβάζει στο Συμβουλίο τα στοιχεία του πληθυσμού που απαιτούνται για την ε, ειδική πλειοψηφία, για την ψηφοφορία ειδική πλειοψηφία και ε, μιλάμε για τα στοιχεία που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στη Eurostat. Όμω ε, υπάρχουν προβλήματα συγκρισιμότητα των δεδομένων έχουμε προβλήματα διπλής ε, καταμέτρησης. Έτσι λοιπόν, ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να βελτιώσει την ποιότητα και ιδίως τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και να αποφύγουμε το μεγάλο πρόβλημα της διπλής καταμέτρησης που έχουμε σήμερα. Η Κομισιόν σε σχέση με το άρθρο 4 θα ήθελε να τονίσει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το άρθρο 4 στον κανονισμό αυτό ή να μην αφαιρεθεί η αναφορά στην ψηφοριδική πλειοψηφία γιατί ε, αν διατηρήσουμε τα βασικά δημογραφικά δεδομένα και τα δεδομένα του πληθυσμού που πετούνται για την ψηφοφορία ειδική πλειοψηφίας είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο έχουμε συγκρίσιμες πληροφορίες ε, για την ειδική πλειοψηφία, αλλά και θα χρησιμοποιείται και οι ίδιες πηγές για δημογραφικές στατιστικές γενικά και για την ψηφοφορία ειδική πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν, επιμένει η Κομισιόν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το άρθρο 4 ελαφρά αναδιατυπωμένο διατυπωμένο ίσως, αλλά θέλουμε να διατηρηθεί αυτή η αναφορά στην ειδική πλειοψηφία στον ίδιο κανονισμό όπως για τις δημοκρατικές στατιστικές γενικά. Επίσης η Κομισιόν θα ήθελε να επιμείνει στο εξή ότι οι διεθνείς συστάσεις ε, τηρούνται, ακολουθούνται κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του πληθυσμού τη χρήση της σύσταση, της συνήθως κατοικίας που βασίζεται στο κριτήριο των 12 μηνών που είναι μια διεθνή σύσταση και που αποφεύγει, μας κάνει να αποφεύγουμε το πρόβλημα της διπλής καταμέτρησης. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό για την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να κλείσω αυτό το σημείο της ημέρης της διάταξης. Και σας υπενθυμίζω όσα υπόθηκαν. Ε, θα θέλαμε να βρούμε έναν συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αν μπορείτε να εργαστείτε απόψε. Αύριο το πρωί, με την συνεδρία των συντονιστών, αφού ολοκληρωθεί η συνεδρία, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε στις 10. Διαφορετικά θα πρέπει να αναστείλουμε και πάλι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 5 που προβλέπει η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Ο εισηγητής είναι ο συνάδελφος Ράνιντελ και θα του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει, να σχολιάσει μάλλον τις τέσσερις τροπολογίες που παρουσιάστηκαν από τον κύριο Νταφ και να μας πει αν υπάρχουν συμβαστικέ τροπολογίες. Ο κύριος Ράντζελ. Ευχαριστώ. Eu devo dizer... Βασικά να σας πω ότι έχουμε τέσσερις ε, τροπολογίες, όλες από τον κύριο Νταφ. Εγώ θεωρώ ότι δύο μπορούμε να τις δεκτούμε όσα έχουν. Έτσι λοιπόν ε, θεωρώ ότι είναι σκόπιμες οι παρατηρήσεις αυτές κυρίως ε, αυτό που σχετίζεται με την εξέλιξη του σημείου 6 και το σημείο 7, το σημείο 6 έχει να κάνει με την Ολομέλεια και το 7 με την δυνατότητα να προετοιμάζεται ένα έγγραφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αρχή καθευθείας που θα παρουσιάζει τις πολιτικές προτεραιότητες για το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Ντάφ επί της ουσίας θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διακυβευτεί η αρχή ε, της ισορροπίας των εξουσιών. Ε, έτσι λοιπόν ε, το Κοινοβούλιο... Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η ιδέα αυτών των δύο τροπολογιών είναι θετική ιδέα. Η ιδέα ότι εμείς πρέπει να έχουμε πραγματική εκτελεστική εξουσία σε ό,τι φορά την οικονομική πολιτική και το Κοινοβούλιο πρέπει όχι μόνο, όχι να είναι αυτό που χαράσει την οικονομική πολιτική, αλλά να ελέγχει την οικονομική πολιτική, δηλαδή να προβαίνει σε έναν έλεγχο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δεκτούμε αυτές τις δύο τροπολογίες που είναι θετικές και το ίδιο θα έλεγα ότι το ίδιο ισχύει για την τροπολογία που προτείνει να διαγραφεί το δεύτερο σημείο του σημείου 16 που είναι η παροχή πληροφόρηση στους βουλευτές. Γιατί όταν μιλάμε για την ενημέρωση των βουλευτών αυτό που διακυβεύεται είναι ότι ξέρετε είχαμε και μια γνωμοδότηση ΑΦΚΟ πέρσι και δεν υπάρχει εδώ καμία καινοτομία. Έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση. Τώρα, στην άλλη τροπολογία που έχει να κάνει με τη διοργανική συμφωνία που διαγράφει, καταργεί το σημείο 17, εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον εκτίματα, τουλάχιστον όσο δεν υπάρχει πραγματική εκτελεστική εξουσία για την οικονομική πολιτική μια πραγματική οικονομική κυβέρνηση, κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ νομίζω ότι υπάρχει νόημα να έχουμε μια διοργανική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου, έτσι ώστε ο δημοκρατικός έλεγχος ε, της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μπορεί να ελοποιείται. Εγώ νομίζω ότι ε, εδώ δεν θα χαίνομαι να το αποσύρουμε όταν γνωρίσουμε ότι ε, η ιδέα αυτή έχει ήδη εκφραστεί και από την ΕΚΟΝ και από την Κομισιόν. Βέβαια, εγώ θα συμφωνούσα με τη θέση του κυρίου Νταφ αν εμείς είχαμε προχωρήσει περισσότερο, δηλαδή αν είχαμε πραγματική οικονομική κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είχαμε και εκτελεστικέ βάσει. Δεν θα χρειαζόμασταν αυτέ τι διευκρινήσει για αυτή τη συμφωνία. Ενώ τώρα όταν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εν εξελίξη, σε μια διαδικασία που δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα, εγώ νομίζω ότι μια διοργανική συμφωνία προσφέρει μια σταθερότητα και βλέπουμε μέσα σε ποιο πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε, επομένω πρέπει να το επιζητήσουμε. Έτσι λοιπόν, εγώ θα δεχτώ, χωρί ε, Τίποτα άλλο. Θα δεχόμουν τις δύο τροπολογίες που προτείνονται για το σημείο 6 και για το σημείο 7 από τον κύριο Νταφ και δεν θα δεχόμουν, δεν θα υπήρχε δηλαδή καμία τροπολο... καμία, κανένα συμβιβασμό για τις προτάσεις που γίνονται για τη διαγραφή του δεύτερου σημείου του σημείου 16 και το σημείο 17 σε σχέση με τη διοργανική συμφωνία. Βεβαίως ε, είμαι διαθέσιμος ε, εδώ για να ακούσω του συναδέλφους, αλλά αυτή είναι η αρχική μου θέση. Βέβαια, αν ακούσω πιστικά επιχείρηματα, μπορεί και να αλλάξω την απόψή μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσσερ Σμίτ έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί τη ευκαιρία θα μιλήσω και τη μετρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για την ενδιαφέρουσα αυτή γνωμοδότηση. Τώρα εγώ δεν θέλω βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπλέκεται στην οικονομική πολιτική των κρατών μελών, αλλά αντιλαμβάνομαι το ότι ε, λέει η συνθήκη και αυτά τα οποία έχει καταθέσει ως τροπολογίες ο κ. Ντάφ, ειδικά στο σημείο 6, είναι πολύ ενδιαφέροντα και λογικά δεν είναι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τα Εθνικά Κοινοβούλια, αυτά τα οποία έχουν την αρμοδιότητα για την πολιτική της ανάπτυξη. Θα ήθελα να σχολιάσω επίσης το σημείο 10, το οποίο τονίζει τον ρόλο των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων και όταν ε, υιοθετηθεί σε κάνα έκθεση και πάει στην Ολομέλεια θα ήθελα να δούμε το που θα γίνει η συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια. Κατά κανόνα βεβαίως όταν μία έκθεση περνάμε στην επόμενη, αλλά νομίζω πως ε, θα έπρεπε εδώ πέρα να δούμε αν πρέπει να προσκαλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα εθνικούς βουλευτές εδώ πέρα για να δούμε ακριβώς το σημείο 10. Νομίζω το σημείο 10 είναι πυρήνα τη συζήτηση που πρέπει να γίνει για την αναπτυξιακή πολιτική στο μέλλον. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια και τον κύριο Ντάφ. Κύριος Ντάφ. Ευχαριστώ. Ναι, οπωσδήποτε συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Ότι πρέπει δηλαδή να δούμε πιο σοβαρά το πώς ακριβώς ε, θα διαρθρωθεί αυτή η συνεργασία μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων για την οικονομική πολιτική της Ένωσης. Και ειδικά για το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου που είναι βεβαίως ένα θέμα το οποίο τα κανονικά είναι αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων και όχι απλά των οικονομικών. Τα συνταγματικά χαρακτηριστικά του πώς οργανώνεται η συνεργασία μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ε, συζήτησης. Ευχαριστώ και τον ε, Παύλο Ράντσελ που αποδέχτηκε τις ε, πρώτες δύο τροπολογίες. Δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να σεβόμαστε την διάκριση των εξουσιών και την εντολή της ε, Κομισιόν, αλλά νομίζω πως στην πράξη νομίζω πως ε, αυτό το οποίο μας ζητάει ο Παύλο εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και άρα νομίζω καλύτερα να μην γίνει και τροπολογία. 3. Προτείνω τη διαγραφή του δεύτερου μέρους του παραγράφου, γιατί αυτή η διάταξη περιλαμβάνεται στην ε, συμφωνία πλαίσιο. δεν έχω καμία αντίρρηση να συμπεριληφθεί, οπότε ευχαρίστως να αποσύρω την τροπολογία 3. Για την τέταρτη τροπολογία για την ε, διοργανική συμφωνία αντιλαμβάνομαι πως είναι της μοδός το Κοινοβούλιο να προτείνει συνεχώς ε, την διατύπωση πιο ε, επισήμων συμφωνιών με την Κομισιόν. Αλλά νομίζω πως είναι ένας δυσκίνητος τρόπος ε, συνεργασίας με την Κομισιόν. Χρειάζεται χρόνος για τις διαπραγματεύσεις. Χρόνος που θα μπορούσε πιο αποτελεσματικά να χρησιμοποιηθεί στην εξέταση της ουσίας της, ε, του, της πολιτικής ε, σταθερότητας και ανάπτυξης των 27 ε, κυβερνήσεων και της Κομισιόν. Και δεν νομίζω πως σε αυτή τη φάση τη μεταβατική ε, μεταβατική φάση της ε, δημοσιονομικής και φορολογικής ολοκλήρωσης να χρειάζεται να επινοήσουμε νέα μέσα. Εγώ ο ίδιος θα προτιμούσα να ενσχοληθεί με αυτά τα ζητήματα η διάσκεψη του 2015 τα ζητήματα δηλαδή οικονομικής διακυβέρνησης και εκεί πέρα ακριβώς θα βρει την φυσική του θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκερέρο. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων. Εγώ θα υπερασπιστώ τη θέση που εκφράζει ο κύριος ε, Ραντζέλ στο σχέδιο γνωμοδότησής του, διότι θεωρώ ότι διέπεται από την επιθυμία να ενισχύσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδίως σε μια χρονική στιγμή όπου οι μεταρρυθμίσεις σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης και ο οποιαδήποτε παρέκκληση διακυβερνητικής φύσεως αυτής τη μορφή της μεταρρυθμίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαχωρισμό και αποδυνάμεση του Κοινοβουλίου όσον αφορά στον έλεγχο αυτό των ε, καινοτομιών που θα έχουμε σε, σαν συνέπεια της οικονομικής διακυβέρνησης. Κατανοώ τους λόγους που οδηγούν τον κύριο Νταφ ε, να παρουσιάσει αυτές τις τέσσερις τροπολογίους. Ε, καταλαώ και τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Ρανχέλ δέχεται τις δύο πρώτες τροπολογίες. Αλλά εγώ φρονώ ότι στην ουσία, εάν ερμηνεύσουμε το κείμενο της γνωμοδότησης του κυρίου Ρανχέλ, που το πνεύμα στο οποίο θεωρώ ότι έχει δομηθεί, ε, θεωρώ ότι αυτό σημαίνει ότι η τροπολογία 1 στην παράγραφο 6 ουσιαστικά λέει ότι το Κοινοβούλιο ανα πάσα στιγμή μπορεί να εκφράσει την άποψή του για τις οικονομικές προτεραιότητες και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αρκεί να υπάρχει μια συμφωνία στη διάσκεψη των Προέδρων και ε, φτάνει στην Ολομέλεια κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι όσον αφορά την άλλη τροπολογία που δεχτήκατε, που ουσιαστικά διαγράφει ε, το κείμενο, αυτό που λέει είναι ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει την εσωτερική του συνένεση για τις πολιτικές προτεραιότητες στην αρχή της θητείας. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δυνατότητα της πολιτικής ε, διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι απλώ η δυνατότητα να δοθεί και ένας πολιτικός προσανατολισμό από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, η οποία δεν θα είναι και απαραίτητο αντίθετη στη θέση τη Κομισιόν. Ε, τα, οι υπόλοιπε δεν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικέ. ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το ίδιο υπερασπιζόμαστε και ε, το ίδιο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων λόγω της ανάγκης βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης και είναι καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και στον έλεγχο των επιπτώσεων που θα έχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην καθημερινή ζωή και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να βρούμε απλώς τους μηχανισμούς προκειμένου να μπορεί να εκφράσει και τη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζουμε μια γνωμοδότηση και η αρμόδια επί της επιτροπής, η Επιτροπή Οικονομισματικών και, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων θα αποφασίσει. Εγώ ως ε, ε, μέλος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα καταψηφίζω τις τροπολογίες αλλά καταλαβαίνω για ποιο σκοπό παρουσιάζονται και κατανοώ και για ποιο λόγο δέχεται τις δύο τροπολογίες ο κ. Ραχέλη. Να δώσουμε λοιπόν τον λόγο στον κύριο Ρανκέ. <coughs> Ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μίλησαν, τον κύριο Μέσσερ, Σμιτ, Νταφ και Γκερέρο. Και να συγχαρώ τον ε, κύριο Γκερέρο, γιατί πραγματικά απέτυχε κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο. Ε, συμφωνεί μαζί μου περισσότερο από όσο συμφωνώ κι εγώ. Θα ήθελα μόνο να πω κάποια πράγματα στον κύριο Νταφ για την τελευταία του παρατήρηση για την διοργανική συμφωνία. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό το οποίο λέει, αλλά θεωρώ επίσης πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε κάποια πίεση της και στο Συμβούλιο. Και αν δεν έχουμε αυτό το, το πλαίσιο, ε, υπομορφή δηλαδή μια διοργανική συμφωνία, θα είμαστε σε μια θέση εξασθενημένη. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να ασκούμε αυτή την πίεση. Εάν με ρωτήσετε το τι θα προτιμούσα, οπωσδήποτε θα προτιμούσα ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων Ε, στο μέλλον. Αλλά ακριβώς επειδή σχεδιάζουμε ένα νέο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε κάποια πίεση και να πούμε ότι εντάξει εάν δεν ε, ε, κάνετε τίποτα θα γίνει μια διοργανική συμφωνία για το ζήτημα αυτό. Για μια στρατηγική, τακτική θέση αλλά Βεβαίω τα συνταγματικά ζητήματα αφορούν και την τακτική και τη στρατηγική των θεσμικών οργάνων. Οπότε θα διατηρήσω τη θέση μου, θα δεχτώ τις δύο πρώτε τροπολογίες και θα απορρίψω τις άλλες δύο. Καλώς. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι περατώθηκε αυτή η συζήτηση για τη γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα ψηφίσουμε στις 5 σήμερα τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο που έχουμε στο υπαρθμό 6 καθεστώς και χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων. Η κυρία Γιαννάκου είναι η συγγήτρια. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είχαμε την 17η Ιανουαρίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας τις τροπολογίες, αλλά μόνο στην αρχική γλώσσα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Γιαννάκου και κατόπιν μπορεί να παρέμβουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η ψηφοφορία θα γίνει πριν από τις 19 Φεβρουαρίου. Κύριε Γιαννάκου, έχετε το λόγο. Ε, υπάρχουν 370 τροπολογίες για την έκθεση. Γεγονός που με εκπλήσει για να είμαι ειλικρινής Δηλαδή υπάρχει πλήθος τροπολογιών από συναδέλφου που ενώ είχαμε συζητήσει πολλές φορές την έκθεση στην Επιτροπή ποτέ δεν εξέφρασαν τις απόψεις αυτές. Και ομολογώ ότι είναι μια δυσάρεστη έκπληξη διότι σας θυμίζω ότι στην πρώτη έκθεση καταρχήν στην οποία κάναμε τις προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρχαν 18 μόνο τροπολογίες στην Ολομέλεια οι οποίες απερίφθησαν όλες και δεύτερον διότι επανειλημμένα συζητήσαμε εδώ για τα πολιτικά κόμματα και οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει τροπολογίες που εκφεύγουν τελείως τις πρότασεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχουν καμία σχέση, δεν μίλησαν ποτέ γι' αυτό. Ούτε πήραν θέση, ούτε εξέφρασαν κάποια άποψη αν λάβουμε υπόψη μας ότι τον Ιούλιο η ιστορία αυτή πρέπει να έχει τελειώσει αν θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσία στα κόμματα και να μπορέσουμε να πάμε στις εκλογές του 2014 με κόμματα με πραγματικό στάτους γιατί αυτό θα τους δώσει και τη δυνατότητα πιθανόν να προτείνουν υποψηφίους για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ. Αντιλαμβανόμεθα ότι με μια τέτοια διαδικασία τα πράγματα δυσκολεύουν να λάβουμε υπόψη μας ότι θα χρειαστεί και πάλι τρίλογος και με το Συμβούλιο. Διότι με την Επιτροπή έχουμε συνεννοηθεί το Συμβούλιο, ορισμένες χώρες του Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι ετώνησα από την αρχή ότι δεν ζητάμε περισσότερα χρήματα, δεν ζητάμε καθόλου περισσότερα χρήματα, ε, έχουν κάποιους φόβους. Επίσης πρέπει να σημειώσω ότι η σοσιαλιστική ομάδα στις τροπολογίες που έχει κάνει μάλλον έρχεται σε καλύτερη συνάφεια με την έκθεση. Αντίθετα, οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και άλλοι συνάδελφοι έχουν κάνει τροπολογίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πρόταση ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε τη δική μου. Αυτό θα δυσκολέψει τα πράγματα κύριε Πρόεδρε ε, βεβαίως θα γίνουν όλα τα αναγκαία. Θα γίνουν δηλαδή συνεννοήσεις με τους Σάντοβου εισηγητές, με τους οποίους ήδη είχαμε βέβαια μία συνάντηση πριν γίνουν οι τροπολογίες και με τη γραμματεία θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά πρέπει να σας πω, ε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ε, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητα ως προς τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, ενώ το Κοινοβούλιο χρηματοδοτεί, και ότι οι αρμοδιότητες όλες πρέπει να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το, αυτή η άποψη, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι τελείως αντιδημοκρατική, διότι δεν είναι δυνατόν τα κόμματα να μην εγγράφονται στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτελεστικό ρόλο, δεν έχει καμιά σε καμία χώρα τα κόμματα δεν εγγράφονται σε υπουργείο ή σε κυβέρνηση. Εγγράφονται στα κοινοβούλια. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι έχω μια πολύ σοβαρή απορία πού βρέθηκαν αυτές οι απόψεις ενώ έχουμε συζητήσει τόσες φορές και πώς ξεφύτρωσαν ξαφνικά όλα αυτά τα οποία θα, διο θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, τη συνεννόηση μεταξύ των τριών οργάνων. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να μας εξηγήσουν, δηλαδή, από πού ξαφνικά μετά από τόσο καιρό συζήτησης ήρθε η έμπνευση να γίνουν τροπολογίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη γραμμή της έκθεσης την οποία γραμμή την είχαμε συναποφασίσει εδώ μέσα και στην πρώτη έκθεση και τώρα. Βεβαίως εγώ θα προσπαθήσω αλλά πρέπει να σας πω ότι η πλειοψηφία των τροπολογιών βρίσκεται τελείως εκτός πραγματικότητας τη της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής μου και δεν είναι αποδεκτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς έχει ζητήσει πρώτα στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει και για το σχέδιο έκθεσης και συμφωνώ πως ε, υπήρξαν πραγματικά αρκετές ε, συζητήσεις αλλά νομίζω πως είναι και λογικό ε, εντός των πολιτικών κομμάτων να ε, έχει ξεκινήσει μια σχετική και έντονη συζήτηση. Οπότε νομίζω πως είναι απολύτως ε, λογικό το ότι τώρα στο διαδικασία της ε, οργάνωσης ενός συμβασμού να καταδεθούν κάποιες τροπολογίες. Ε, και εγώ ίδιος υπέβαλα κάποιες ε, τροπολογίες ε, για την ομάδα μας που είναι στη γραμμή της μέχρι τώρα τοποθέτησής μας για τον οργανισμό αυτόν. Και πρώτον να σκεφτούμε δηλαδή γενικά πού πρέπει να έχουν έδρα αν θέλετε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τι θέση έχουν και είχαμε και συζητήσεις με τον Επιτροπό για αυτό το θέμα και συζητήσαμε το ότι η Κομισιόν αφενός λέει ναι, θέλουμε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν έναν μεγαλύτερο, πιο κυρίαρχο ρόλο, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνουν στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου στη χώρα όπου έχουν εγγραφεί. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα Δηλαδή δεν θα είναι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κόμματα αυτά. Εμείς λέμε πως θα πρέπει να, είναι, να έχουν μια αντιμετώπιση ανάλογη με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εξαρτήτως του που έχουν εγγραφεί και να είναι μια κατηγορία σου εγγένερης στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών και του δικαιώματος ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, του δικαιώματο ε, του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε. Θα ήθελα επίσης να πω το δεύτερο, τη δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια αποπολιτικοποίηση της διαδικασίας αυτής της εγγραφής. Δηλαδή, οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να ιδρύσουν ένα τέτοιο πολιτικό κόμμα έχουν έναν συγκεκριμένο ρόλο. Και έχουν τα δικαιώματα. Δηλαδή, όπως και σε πολλά κράτη-μέλη, εγγράφονται σε έναν κατάλογο, σε ένα μητρό τα πολιτικά κόμματα και ε, αυτό είναι μια διοικητική διαδικασία, όχι μια πολιτική αξιολόγηση. Αυτή έρχεται μετά από τη δραστηριότητα του πολιτικού κόμματος, αν υπάρξουν αμφιβολίες κτλ. Οπότε εμεί θέλουμε να υπάρχει έτσι όπως είπα αυτή η διαδικασία. Τρίτο θέμα και τέτοια κατηγορία τροπολογιών που έχουμε καταθέσει και νομίζω πως εδώ πέρα θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή θέση γιατί η συζήτηση στο παρελθόν αυτό έχει ρίξει το πώς πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ μεγάλων και μικρών παλαιότερων και νέων πολιτικών, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που θα πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες παρέμβασης στην πολιτική συζήτηση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα ε, εξού και η πρότασή μας να παραμείνουμε στο τωρινό επίπεδο της ε, χρηματοδότησης, δηλαδή 15% και 85% όσον αφορά την, την κατηγοριοποίηση όσον αφορά δηλαδή τον, τον αριθμό των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η συζήτηση για το πού πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο δημοκρατική είναι, σε ποιο βαθμό μπορούν οι πολίτες ε, να παρέμβουν στην ε, λήψη των ε, αποφάσεων κλπ. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει μέσω της ισότιμης δυνατότητας παρέμβασης των κομμάτων. Και τέταρτον, από πότε, από ποια στιγμή έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Είναι έβδομο των καρτών μελών, είναι πέμπτο, είναι το ένα τέταρτο. Εμείς θεωρούμε, όπως είπαμε και για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, πως πρέπει να είναι χαμηλό το κατόφλι αλλά και αντιπροσωπευτικό. Γι' αυτό προτείνουμε το ένα πέμπτο των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. από το οποίο θα προέρχονται τα κόμματα τα οποία θα φτιάξουν ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος θα έχει το λόγο. Ehm. Ευχαριστώ. Η συνεδρία, στην συνεδρίαση των ε, σκιωδών εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συζήτηση την οποία θα ήθελα να αναφέρω γιατί συζητήσαμε ζητήματα δημοκρατικής νομοποίησης σε πολλά επίπεδα. Ότι δηλαδή το μοντέλο το οποίο έχουμε όπου υπάρχουν βουλευτές που αποφασίζουν σε ποιο βαθμό τα, τα κόμματα μπορούν να ανταποκριθούν ε, στις απαιτήσεις αυτές ε, είναι ένα πρόβλημα. Βεβαίως ε, εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω βεβαίως κανένα συνάδελφο αλλά κόμματα τα οποία δεν δέχονται τις δημοκρατικές αξίες και τα δικαιώματα κτλ. Ε, τι, θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εάν ε, εκλέξει κάποιου εκπροσώπου οι οποίοι μετά απορριφθούν. Εάν δηλαδή είναι κάποιο ένα νέο κόμμα και απορριφθεί από του υπόλοιπου, έχουμε ένα πρόβλημα. Ξέρω πως ο κύριος Ντάφ έχει καταθέσει μια σχετική τροπολογία την οποία θα ε, στήριζα. Το κομμάτι αυτό της έκθεσης που έχουμε τώρα δημιουργεί τεράστια προβλήματα όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης των κομμάτων. Βεβαίως πρέπει να έχουμε μια έγκριση των νέων κομμάτων γιατί μιλάμε και για πρόσβαση και σε πολλά λεφτά και δεν είναι λογικό και δεν είναι και προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνουν αυτό τον έλεγχο οι βουλευτές. Ε, κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει. Και αυτό είναι και προς το συμφέρον των βουλευτών για να μην μπορεί κανείς ε, να τους ε, κατηγορήσει ότι προσπαθούν να εμποδίσουν νέους αντιπάλους και ανταγωνιστές. Νομίζω πως αυτό το στοιχείο πρέπει να βγει από την έκθεση και να ξαναγραφτεί. Αλλιώς είμαστε μετά ανοιχτοί σε επιθέσεις και θα νομοποιηθούν μετά κάποια κόμματα τα οποία δεν θα θέλαμε να δούμε ως δημοκρατικά εκλεγμένα κόμματα. Ωραία. Κύριε το λόγο. Δεν νομίζω Ε, πως ε, η κυρία Γιαννάκου πρέπει να, να από τον αριθμό των τροπολογίων. Ξέρουμε πως είναι επίμαχο το ζήτημα. Διαφέρουν οι πρακτικές ε, από χώρα σε χώρα. για τη δομή και την ρύθμιση και τον τόνο που έχει νομοθεσία περί πολιτικών κομμάτων. Και σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, η εκτελεστική εξουσία είναι αρμόδια για την εγγραφή πολιτικών κομμάτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη, ε, έτσι συμβαίνει. Και βεβαίω ε, θα δούμε και διαφωνίες ε, στο Συμβούλιο, οι οποίες αντιλαμβάνουμε πως είναι μεγάλες. Και θα πρέπει να υπάρξει τριμερής διάλογος πριν ε, καταλήξουμε κάπου με αυτή την νομοθεσία. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το χρειαζόμαστε αυτό είναι λόγω της κακής ποιότητας της διατύπωσης της Κομισιόν. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη ορισμοί των ε, των μελών του κανονισμό δηλαδή δεν είναι σαφές το τι, τι θέλουν να πούνε εδώ πέρα μιλάνε για το να είναι ένα άτομο μέλος ενός κόμματος ή μιλάνε για τα για τους βουλευτές και τα, και τα γραφεία επίσης του κόμματος. Και εδώ πέρα χρειάζονται διευκρινήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Σόλτς πως πρέπει και το έχω ξαναπεί αυτό να βρεθεί ένας τρόπος εγγραφής ε, ελέγχου που θα είναι αυστηρός, ε, αντικειμενικός και ως το δυνατόν πιο αμερόληπτος. Η προτιμησή μου προσωπικά είναι μία εκλογική επιτροπή, μία αρχή η οποία θα ε, είναι κάπως ανεξάρτητη από την Κομισιόν. Αλλά η λεγόμενη Επιτροπή Σοφών είναι μάλλον μια επαρκής ε, δικλίδα ασφαλείας. Το δέχομαι λοιπόν, αλλά θα ήθελα να αυξηθούν τα μέλη από 3 σε 9. τρία μέλη που θα ορίζουν τα τρία θεσμικά όργανα. Επίσης, θα ήθελα να εισαχθεί η ιδέα πως ε, κυρώσεις ε, και ποινές ε, πρέπει να γίνονται μέσω πράξεων καταξιοδότηση. Πρέπει να πούμε επίσης ξεκάθαρα το τι είναι ένα πολιτικό κόμμα. Δεν είναι απλά μια, ένα σύνδεσμος ανθρώπων με ίδιες πολιτικές ιδέες ε, είναι ένας μηχανισμός εξτρατιών με στόχο την κατάκτηση της εξουσίας εδρών και ψήφων. Και όπως είπα στο παρελθόν, δεν ναι, θεωρώ πως η Κομισιόν έχει αντιληφθεί το σε τι χρησιμεύουν τα πολιτικά κόμματα. Και το τι νέες ευθύνες θα έχουν. Τέταρτο. Για το ζήτημα των ορίων. Εμείς το συζητήσαμε στην ομάδα μας και καταλήξαμε πως για να διασφαλίσουμε πως ε, τα πολιτικά αυτά κόμματα θα είναι όντως διεθνή πρέπει να ορίσουμε το κατόφλι στο 1 τρίτο των κρατών μελών. και των εθνικοτήτων σε ένα πολιτικό κόμμα. Επίσης έχει μπει μια ρήτρα για να μην υπάρχει διπλή καταμέτρηση. και για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια της ε, διαδικασίας αυτής ε, της ε, εγγραφής που θα πρέπει της διαδικασίας τεκμηρίωσης που θα πρέπει να δημοσιεύσει το Κοινοβούλιο ε, ως ε, μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Νομίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία επί αυτών και αναμένω και την περαιτέρω συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε κύριε Ντάφ. Ο κύριος ε, Ραντσέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Μαριέτα Γιαννάκου για το έργο της και βλέπω ότι θα έχει πολύ περισσότερη δουλειά με όλες αυτές τις προτάσεις τροπολογιών. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τη Μαριάτα κατά κάποιο τρόπο, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες. Δηλαδή, συμφωνώ ότι είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει επί μακρόν, αλλά είναι προφανές ότι είναι τόσο θεμελιώδες που είναι λογικό στο στάδιο αυτό και επειδή είναι το κρίσιμο στάδιο μάλιστα, να υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Αν και θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί είμαι ένας από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν πάρα πολύ εντατικά αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν είχαν πάρει το λόγο προηγουμένω. Δεν είχα συζητήσει με τη Μαριέτα για την τελική μου θέση. Ακόμη και αν είχα μια θέση από την αρχή. Πρέπει να πω λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ το Κοινοβούλιο να έχει εδώ αρμοδιότητα εγγραφής. Αυτή είναι η δική μου θέση όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργήσει υποψία ότι τα κόμματα που είναι ήδη στο Κοινοβούλιο κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να επηρεάσουν ή να ελέγξουν τα κόμματα που θα δημιουργηθούν στα κράτη-μέλη. Αυτή ήταν πάντοτε η θέση μου και πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες όπου το Κοινοβούλιο δεν ε, έχει επιρροή. Παραδείγματο χάρη στην περίπτωση τη Πορτογαλία, αρμόδιο είναι το συνταγματικό δικαστήριο. Δηλαδή, ε, ούτε καν ε, η δίκηση που υπάρχει δεν είναι αρμόδια για την εγγραφή των κομμάτων. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να έχουμε ένα εξαρτητό φορέα φυσικά. Εγώ πιστεύω και πιθανότητα αυτό θα είναι ένα συνδεσμό ότι είναι δυνατό να έχουμε μια ανεξάρτητη διοίκηση εντό του Κοινοβουλίου. Δηλαδή θα είναι δυνατό να έχουμε ένα φορέα που θα είναι υπεύθυνο για αυτά τα εκλογικά θέματα και για θέματα που αφορούν τα κόμματα και θα υπάρχει στους κόλπους του Κοινοβουλίου. Θα είναι ανεξάρτητος με αυτός ο φορέας, αλλά θα είναι εντό των κόλπων του Κοινοβουλίου. Είναι δυνατόν. Αυτό και εγώ θα το δεκόμουν αυτό εύκολα. Όμως, να πω ότι με ανησυχεί αυτό το ζήτημα. Και αποτελεί ανησυχία όχι μόνο γιατί θεωρητικά Είναι δύσκολο να δεκτούμε αυτό, να γίνει δεκτό αυτό τουλάχιστον σε κάποιες χώρες ε, και γι' αυτό το αντιμετωπίζει και το Συμβούλιο έτσι αυτό το ζήτημα, αλλά γιατί αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που υπάρχει σε κάποιες χώρες ενώ σε άλλες δεν υπάρχει. Δηλαδή ουσιαστική επαλήθευση του προγράμματος του κόμματος ή της δραστηριότητας του κόμματος. Αυτή η ρήτρα ότι θα πρέπει να σέβεται τις δημοκρατικές αξίες, του κράτους δικαίου κτλ. Είναι κάτι ιδιαίτερα αποδεκτό, αλλά είναι και επικίνδυνο ταυτόχρονα. Γιατί τότε ελέγχουμε την ιδεολογία του κόμματος, την ιδεολογία των κομμάτων και θα έλεγα αυτό είναι παράδοξο της δημοκρατίας. Δηλαδή να έχουμε αυτόν τον έλεγχο για να υπερασπίσουμε τη δημοκρατία κατά της δημοκρατίας. Είναι κάπως δύσκολο αυτό το ζήτημα. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα συνταγματικής φιλοσοφίας. Και η δική μου πιο σημαντική τροπολογία πιθανότητα δεν είναι και τόσο επίμαχη και αφορά αυτή την εκλογική διοίκηση. Είναι να προσθέσουμε σε αυτή την ουσιαστική ρήτρα συμβατότητας, δηλαδή να λέμε δημοκρατικές αξίες, αξία του κράτους δικαίου και μια υποχρέωση αμεροληψίας και ουδετερότητα, για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την αρχή του πλουραλισμού. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδέα του, του πλουραλισμού. Ο φορέας που θα έχει αυτόν τον ε, ουσιαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του κόμματο θα πρέπει να έχει την εξή υποχρέωση, να προσπαθεί να πετύχει τόσο δυνατόν μεγαλύτερο πλουραλισμό. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Να δώσουμε στο φορέα ελέγχου, δηλαδή να μην προσπαθήσουμε να έχουμε έναν ιδεολογικό έλεγχο και να αποφαινόμαστε επί της ιδεολογίας, αν είναι καλή όχι. Ξέρω ότι υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, όπου κάποιες ιδεολογίες απαγορεύονται από το Σύνταγμα, το ίδιο συμβαίνει με την Πορτογαλία, αλλά μόνο με τις ε, ακροδεξιές ιδεολογίες, αν είναι αριστερές δεν υπάρχει πρόβλημα, ακόμη και αν μιλάμε για στελινισμό. Αλλά πραγματικά δεν μου αρέσει μια τέτοια είδους παρέμβαση. Τι κατανοώ σε χώρες όπως δικές μου ή τη Γερμανία για ιστορικούς λόγους. Δεν είναι όμως πολύ υγιές ε, για το δημοκρατικό σύστημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντική αυτή η τροπολογία να προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ότι ο ουσιαστικός έλεγχος δεν είναι ιδεολογικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν σαφές για μας, αλλά δεν ήταν σαφές για κάποιους άλλους. και να αναφέρουμε αυτή την αρχή της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και του μέγιστου δυνατού πλουραλισμού. Και στη συνέχεια θα ήθελα ε, να είναι αρμόδια η Επιτροπή, αλλά μπορώ να δεκτώ και άλλες λύσεις. Αλλά αυτό το ζήτημα συζητήθηκε εις βάθος εδώ, θυμάμαι, και άλλους συναδέλφους, τον κύριο Νταφ, τον κύριο Χεφνέρ, τουλάχιστον μπορώ να θυμηθώ ότι είχαν ε, αναφερθεί επί μακρόν σε αυτό το θέμα, δεν είναι νέο το ζήτημα, ούτε θα λυθεί τώρα. Μάλλον ε, είναι η τελευταία δυνατότητα να τα επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι η Μαριέτα όπως πάντα με την ευαισθησία που τη διακρίνει, θα πετύχει ένα πολύ καλό συμβιβασμό που να μπορεί να δώσει στο Κοινοβούλιο μια ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις στις οποίες θα πρέπει να μπούμε με τα υπόλοιπα όργανα. Ευχαριστώ, κύριε Γαζέλ. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι η συγγήτρια δεν ε, μπορεί να παραπονιέται για την ομάδα των σοσιαλιστών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τροπολογιών, καθώς παρουσιάσαμε 14. Και αυτό σημαίνει το 3,47% των τροπολογιών που παρουσιάστηκαν για την έκθεσή σας. Δηλαδή, ήμασταν ε, γενικά υπέρ ε, της γενικής θέσης σας κυρία εισηγήτρια και να θυμηθείτε πόσο μου έκανε να υποφέρω η κυρία Γιαννάκο με το άρθρο 70. Αλλά τέλος πάντων καλά τα πήγαμε τελικά. Πιστεύω ότι κάποιες από τις συζητήσεις ε, που έχουμε είναι σημαντικές. Δηλαδή το ότι η δική μου ομάδα δεν παρουσιάζει μεγάλο αριθμό τροπολογιών δεν σημαίνει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ε, πολλά ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητο να συζητηθούν εδώ για να ενισχύσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ίδια τη Μαριέτα όταν θα διαπραγματευτεί στον τριμερή διάλογο. Γιατί εγώ θεωρώ και νομίζω ότι το ίδιο θεωρεί και η κυρία Γιάννεκο και αναφέρθηκε ο κύριος Ντάφ σε αυτό ότι στο Συμβούλιο, στους κόλπους του Συμβουλίου υπάρχει σύγχυση και υπάρχει γενικά ε, κάποια ε, ουσιαστικά αρνητική στάση. Τώρα, το θέμα που θέτει μεγαλύτερη συζήτηση, το θέμα της εγγραφής του Μητρώου. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να προσδιορίσουμε τα αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή, για το Μητρώο, παρά να λέμε ποια είναι η αρχή που προβαίνει στην εγγραφή. Αν η αρχή που προβαίνει στην εγγραφή ουσιαστικά διέπεται η λειτουργία της από μία σειρά κριτηρίων αδιαμφισβήτητων, τότε δεν έχει σημασία αν θα είναι η Κομισιόν ή αν θα είναι το Κοινοβούλιο. Αν πρόκειται για τον αριθμό των χωρών, την παρουσία των βουλευτών και ε, στα καταστατικά ρητά. Δεν υπάρχει αντίρρηση, ε, δεν καταφέρονται κατά των ανεφισβήτητων αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα δυνατότητα να είναι η Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο νομίζω είναι δευτερεύον ζήτημα. Και θα πω και κάτι ακόμη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλουμε ότι η Κομισιόν μπορεί να είναι ουδέτερη και το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι μεροληπτικό. Δεν ξέρω γιατί το υποθέσαμε αυτό. Μάλιστα πιο πλουραλιστικό είναι το Κοινοβούλιο από την Κομισιόν. Και είναι επομένως πιο δυνατός ο έλεγχος μεταξύ των ε, έλεγχων και των ισορροπιών της εξερμπάλασης μέσα στο Κοινοβούλιο παρά στους κόλπους της Κομισιόν που ουσιαστικά παρουσιάζει κάποιες ε, προκαθορισμένες τάσεις σε σχέση με το Κοινοβούλιο σε κάποιε συνεδριάσει που είχαμε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σκιώδη εισηγητής, αλλά έχω πει ότι δεν είμαι κατά να δημιουργηθεί ένα μονοδοδοτικό συμβούλιο που κατά κάποιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια αρχή, ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο που κατά κάποιο τρόπο να καθορίζει τι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται. Γιατί τελικά όταν υπάρχει μια σύγκρουση και για το αν ένα κόμμα πληρεί ή δεν πληρεί την αρχή του να σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι η πολιτική δομή της Ένωσης, που δεν είναι οι πολιτικές της Ένωσης που μπορεί να καταφέρεται κατά τη ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κατά των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Όταν υπάρχει λοιπόν μία σύγκρουση πάντοτε θα ε, υπάρχουν υποκειμενικά κριτήρια και πάντοτε θα έχουμε ένα δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει απόφαση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Έτσι λοιπόν, Μαριέτα, αν ε, μπορούμε να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες, τόσο το καλύτερο. Αλλά εγώ θεωρώ το σημείο που πρέπει να συζητήσουμε αφορά τη σαφήνεια των αντικειμενικών κριτηρίων, γιατί όταν καθοριστούν τα κριτήρια τότε θα υπάρχει και περιορισμένο περιθώριο ελιγμών. Τώρα, σε σχέση με τις συγκεκριμένε τροπολογίε που παρουσίασε η δική μου ομάδα, πιστεύω ότι οι περισσότερε ε, δεν είναι ιδιαίτερα επίμαχε. Κάποιε έχουν να κάνουν με τη σχέση μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αντίστοιχο κόμμα που ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια, δηλαδή δυνατόν να υπάρχουν και σχετικές δωρεές. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των διοικητικών οργάνων των πολιτικών κομμάτων, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και κάποια άλλα θέματα, κάποιες άλλες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με, τη γενική, με το γενικό σεβασμό γενικών κριτηρίων, παραδείγματο χάρη να υπάρχει ε, ε, εκπροσώπηση και των δύο φύλων. Και Κλείνοντας, να πω το εξή. Πιστεύω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο, γιατί, όπως είπε και η Μαριέτα, αν θέλουμε να έχουμε αυτή την νομοθεσία για το 2014 δεν μπορούμε να διονύζουμε τη συζήτηση εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώ ε, όταν το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει, θα πρέπει να ξεκινήσει και μια πολύπλοκη περίοδος διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Κυρίως γιατί το Συμβούλιο δεν έχει μία ομόφωνη θέση, ούτε μία σαφή θέση στα περισσότερα σημεία. Και πρέπει να επισημάνω ότι παραδόξως, και αυτό είναι ένα παράδοξο κύριε Ραντσέλ γιατί μιλήσατε για το δημοκρατικό παράδοξο, ένα από τα παράδοξα είναι ότι επί τη εθνικά πολιτικά κόμματα δεν θέλουν ε, ε, να έχουν περισσότερη ουσιαστικά σχέση και επιπτώσεις με τις ευρωπαϊκές πολιτικές της οικογένειας. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλές δυσκολίες να προχωρήσουμε στο ιστορικό του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρόνς. Η τροπολογία 3 λέει ότι αρχηγός η Επιτροπής μας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνει πολιτικούς που εκπροσωπούν πολιτικά κόμματα, θα αποφασίζει κατά πόσον κάποια κόμματα προσυπογράφουν κάποιες υποκειμενικές θέσεις. Αυτή είναι κανονικά δικαστική ή μη δικαστική απόφαση που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να λαμβάνεται από δικαστικό σώμα και όχι από μια συνέλευση πολιτικών. Ε, είπαν ότι θα έπρεπε να έχουμε κάποια ενδιάμεση οδό, μια ομάδα σοφών ή πιο πολιτικά ορθό σοφούς ανθρώπους. Εγώ όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να λαμβάνεται η απόφαση από ένα δικαστήριο που ε, δεσμεύεται από νομικέ διαδικασίες και από το κράτος δικαίου. Το άρθρο 9 λέει ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να διασφαλίζουν ισότητα των φύλων ε, και εγώ και κάποιοι άλλοι θα ήθελα να έχουν περισσότερες γυναίκες σε ρετά σώματα παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλύτερα αποτελέσματα από άλλους στο θέμα αυτό. Αλλά το να υπάρχει περιορισμός φύλου θα δημιουργήσει ε, μια σειρά ε, περιορισμών, όπως και οποιοδήποτε άλλος δημογραφικών περιορισμών, θα δημιουργήσει προβλήματα για την άποψη που έχουν κάποιοι για πολιτικά ιδεολογικά ζητήματα και αυτό κατά την άποψή μου είναι περιττή ε, περιττός όρος για να επιβάλλουμε σε ένα πολιτικό κόμμα. Ε, ένα πολιτικό κόμμα θα πρέπει να ε, καθορίζει μόνο του ε, ποιος θα πρέπει να εκλέγεται, διότι αν ε, του πάρουν τη δυνατότητα αυτή δεν είναι πλέον ανεξάρτητο, είναι μόρφωμα του κράτους. Το άρθρο 17 λέει ότι λόγω πολιτικής ερετικής τάσης μπορεί να του αρνηθούμε χρηματοδότηση, αλλά μπορούμε και να το καταργήσουμε το κόμμα αυτό. Εδώ παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερης του συναθρίζεστε. Αν δούμε διάφορα πολιταρχικά καθεστώτα, τα περισσότερα εξ αυτών δεν απαγορεύουν τη δημιουργία άλλων κομμάτων. Αυτό που κάνουν είναι ότι απαγορεύουν τη δημιουργία άλλων κομμάτων χωρίς την άδειά τους. Και αυτό ουσιαστικά προτείνουμε και εμείς εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπρόνς και τώρα ο κύριος Χέφνερ έχει το λόγο. Ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για το ότι μόλις μπήκα σε αυτή την ε, αίθουσα. Ξύπνησε 7 η ώρα σήμερα στο Μόναχο, ήμουν 9 η ώρα στο αεροδρόμιο, αλλά μόλις ε, πριν από 2 ώρες αναχωρήσαμε λόγω του χιονιού και του χάους που επικρατεί στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, καιρικά φαινόμενα που χαλάνε τα σχέδιά μας. Και άρα έχασα το πρώτο μέρος της συζήτησης και ειδικά την παρουσίαση της κυρίας Γιαννάκου. Και ανησυχώ ε, για το ότι κάποια πράγματα τα οποία θα πω έχουν ήδη ίσως ακουστεί. Οπότε δεν μπορώ και να απαντήσω σε πράγματα τα οποία δεν άκουσα, απλά θα παρουσιάσω μόνο τα σημαντικότερα κατά την ε, άποψή μου. Και μετά βεβαίως ε, πάνω σε αυτά έχει καταθέσει και τροπολογίες η ομάδα μου. Πρώτα απ' όλα, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία χρειάζεται ευρωπαϊκά κόμματα. Δεν αρκεί μια ευρωπαϊκή δημοκρατία με εθνικά κόμματα, ούτε αρκεί ε, να υπάρχουν μόνο εθνικά θέματα, εθνικοί υποψήφοι και προεκλογικές εκστρατείες. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρχουν και ευρωπαϊκά θέματα και ευρωπαίοι υποψήφοι και άρα ευρωπαϊκές συζητήσεις και άρα η ύπαρξη ευρωπαϊκών κομμάτων έχει μεγάλη σημασία. Τα ευρωπαϊκά κόμματα ενισχύουν την εκπροσώψη των Ευρωπαίων πολιτών μέσω των εθνικών κομμάτων και έτσι μπορούμε να έχουμε οικογένειες κομμάτων που δεν είναι μόνο εκλογικοί συνασπισμοί αλλά μπορούν να έχουν κάποιες κοινέ ιδέες για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η Ευρώπη για να μπορούν να επιλέγουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτά νομίζω είναι το υπόβαθρο της συζήτησης ε, που κάνουμε τώρα. Και δεύτερον, κάτι που μου φαίνεται πολύ σημαντικό, θεωρώ πως πριν, πριν μπούμε σε λεπτομέρειες πρέπει να συνεννοηθούμε για το τι εννοούμε ε, όταν λέμε κόμμα, τι εικόνα έχουμε για το κόμμα. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως τα κόμματα δεν είναι κάποια κρατικά ή μη κρατικά μορφώματα, αλλά διαμορφώνονται από πολίτες που έχουν κοινέ πολιτικές ιδέες και θέλουν να τις προωθήσουν και άρα συνασπίζονται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί βεβαίως θα διαμορφώσει το νομικό πλαίσιο. Πρέπει να αποφύγουμε ε, το να δώσουμε κάποιο επίσημο κρατικό καθεστώς ε, στα κόμματα και πρέπει αυτό να αντικατοπτρίζεται και στο καθώς και στο καταστατικό αυτό. Και έρχομαι άρα στο ερώτημα το εάν οι απαιτήσει που υπάρχουν για την εγγραφή των κομμάτων αυτών είναι πολύ υψηλές. Ειδικά αν συζητάμε επί τη βάση της δημοκρατίας ε, στις χώρες μας υπάρχουν ε, χώρες που δεν αντιλαμβάνονται το ερώτημα. Τι, τι είπα να πει καταγραφή των κομμάτων. Σε πολλές χώρες δεν αποφασίζει κανείς ε, για κάτι τέτοιο. Απλά αποφασίζουν οι πολίτες ε, να συστήσουν ένα κόμμα και αυτό αρκεί. Αν έχουν επαρκή μέλη και ένα δημοκρατικό καταστατικό, ένα προεδρείο κτλ. Περισσότερα χρειάζονται βέβαια για τη συμμετοχή στις εκλογές. Ε, εκεί πέρα θα πρέπει να υφίσταται οργανωτικά ε, και να εκπροσωπείται σε κάποιες χώρες ε, το κόμμα και ακόμη ψηλότερες πρέπει να είναι οι διατάξει για τη χρηματοδότηση. Γιατί η χρηματοδότηση βεβαίω θα εξαρτηθεί από την επιτυχία και θα πρέπει να αυξάνεται όταν περισσότεροι πολίτες ψηφίζουν αυτό το κόμμα και να μειώνεται ή να καταργείται όταν ε, ε λίγοι ή ελάχιστοι πολίτες επιλέγουν αυτό το κόμμα. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ πως είναι λάθος είναι να θέλουμε να τα συνοψίσουμε όλα αυτά σε ένα. Δηλαδή εγγραφή, ε, πρόσβαση στις εκλογές και ε, χρηματοδότηση και μάλιστα με το ίδιο κατόφλι. Γιατί αυτό το οποίο είναι λογικό για τη χρηματοδότηση, δηλαδή η σύνδεση με τον βαθμό επιτυχίας, δημιουργεί, ε, αν το μεταφέρουμε στην εγγραφή, την εντύπωση πως θέλουμε να σχηματίσουμε ένα κλειστό κλαμπ και να εμποδίσουμε ε, νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν θέλουμε. Αντιθέτως πιστεύω πως ο καθένας από εμά, ο οποίος ε, ε, θεωρεί, ε, ο οποίος βλέπει αυτό το ζήτημα, θεωρεί πως πάνω από το δικό του κόμμα βεβαίως σημαντικότερη είναι η δημοκρατία και θα πρέπει να παραμείνει εύκολη η διαδικασία σχηματισμού ενός ε, ευρωπαϊκού κόμματος και να μην ε, είναι ίδια ε, με την χρηματοδότηση. Γι' αυτό θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Επίσης μου μετέφεραν πως δεν είχαν ανακοινωθεί ε, εκ των προτέρων πολλές ε, τροπολογίες. Εγώ το είχα πει ήδη εξ αρχής ε, πως όσους ρώτησα είπαν το ίδιο πράγμα. Γιατί ε, είχα πει κάποια πράγματα, αλλά ίσως δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Επίσης, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής είχε αποτελέσει αντικείμενο συνένεσης ε, και είχαμε συμφωνήσει και στο τωρινό καταστατικό, δηλαδή ότι ένα 15% της συνολικής ε, χρηματοδότησης ε, θα μοιράζεται γενικώ μεταξύ των κομμάτων και το 85% αναλόγως με την εκλογική επιτυχία. Και γιατί είναι αυτό ε, σημαντικό, γιατί τα κόμματα τα οποία θα έχουν αυτό το καστός θα πρέπει να έχουν ε, κάποια ε, έσοδα τα οποία θα διασφαλίζουν μια ελάχιστη λειτουργία, κάποια γραφεία, κάποιους ε, υπαλλήλους. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ και θεωρώ πως ε, ένα 15% είναι ένα λογικό τέτοιο ε, ποσό. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να αναμειωθεί. Εγώ είμαι υπέρ του να παραμείνουμε στο ποσό που έχουμε τώρα. Το τρίτον το ανέφεραν ε, ήδη πολλοί συνάδελφοι το να λάβουμε εμείς την ε, απόφαση ως κοινοβούλιο για το ποιος πρέπει να αναγνωριστεί ως ε, Ευρωπαϊκό Κόμμα είναι κάτι το οποίο θεωρώ κάπως προβληματικό. Δεν είμαι σίγουρος το εάν εμείς που εκπροσωπούμε ήδη κόμματα έχουμε την απαραίτητη ανεξαρτησία. Γι' αυτό θα ήθελα μια διαδικασία σε δύο φάσεις. Μια διαδικασία όπου πρώτα απ' όλα ε, θα υπάρχει μια απόφαση κάποιας αρχής ε, με βάση κάποια τυπικά κριτήρια και μετά με βάση την σύσταση αυτή το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει την ε, απόφασή του και πρότεινα να σχηματιστεί ένα σώμα το οποίο θα αποτελείται από ε, αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις ε, εκλογικές επιτροπές στα κράτη-μέλη. Υπάρχει νομίζω κάτι ανάλογο σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι ήδη αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την εξέταση αυτών των ε, ζητημάτων και με βάση λοιπόν τη δική τους σύσταση θα μπορούμε να αποφασίσουμε. Οπότε θα μπορεί να ε, λαμβάνει την αλλαγή απόφαση χωρίς να σχηματιστεί μια νέα γραφειοκρατία. Και τέλος, για, όσον αφορά τη μεταφορά ετησίων ε, πλεονασμάτων, αυτό δεν αφορά μόνο τα κόμματα, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ιδρύματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να ισχύσει και για τα ιδρύματα. Έχω και κάποια άλλα πράγματα, αλλά ο χρόνος πιέζει. Ε, δύο πράγματα θα ήθελα να πω ακόμα. Πρώτον, έχω την εντύπωση πως δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αν ε, λάβουμε υπόψη, που υπάρχουν, αν λάβουμε τις προθεσμίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για την προετοιμασία των εκλογών, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, ε, και όπου πρέπει να αλλάξει ο νόμος αν είναι να λάβουν υπόψη αυτές τις προθεσμίες θα πρέπει μέχρι το καλοκαίρι το αργότερο να καταλήξουμε σε μία απόφαση και δεύτερον έχουμε πολλές ε, τροπολογίες και εγώ θεωρώ πως με βάση αυτές τις ε, τροπολογίες μπορούμε να συνεργαστούμε οι κοινοβουλευτικέ ομάδες ε, με την εισηγήτρια και με τους κοιοδησηγητές για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμών για να μειωθεί και ο αριθμός και να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ θέσεις. Για να πάμε μετά και στη διαπραγμάτευση με Συμβούλιο και Κομισιόν. Τέλος, ε, ευχαριστώ την ε, κυρία Γιαννάκου για την πολύ δύσκολη αυτή έκθεση και για τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά της. Θεωρώ πως θα καταλήξουμε νομίζω και σε ένα καλό αποτέλεσμα να συνεχίσουμε έτσι σε αυτή την επικοδομητική ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ κύριος Βίλαντ. Ε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρως με αυτά τα οποία είπε ο κ. Σέφνερ και εγώ ε, ήρθα αργά λόγω των συνθήκων. Ελπίζω να μην επαναλάβω πολλά πράγματα. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος. Δηλαδή, πριν από ένα έτος είχα πει ε, τα βασικά πράγματα τα οποία υπάρχουν στην ε, τοποθέτησή μου. Δεν δηλαδή, αντιλαμβάνομαι λοιπόν πού είναι το, το πρόβλημα. Τέλος δεν θα μπω τώρα στις ε, λεπτομέρειες. έχω καταθέσει κάποιε τροπολογίες όσον αφορά του ορισμού Πρώτον, για τον διαχωρισμό κόμματο, εκλογών και χρημάτων. Συμφωνώ κάπως με τον κύριο Χέφνερ. Πρέπει να γίνει εύκολο ή ευκολότερο, εν πάση περιπτώσει, ε, να αναγνωριστεί ένα κόμμα ως Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα και να μπορεί να κατέβει και στις εθνικές εκλογές αλλά βεβαίως ε, έτσι θα μπορούν παραδείγματο χάρη κάποια κόμματα να έχουν 1-2-3% κάποιου λίγου βουλευτέ και να συνεισφέρουν παρόλα αυτά. Δεύτερον, όσον αφορά τα, τα χρηματικά, εγώ θα ήθελα έναν ε, διαχωρισμό για να ξεπεράσουμε αυτή τη διαμάχη 15-85 ή 10-90 ή 20-80. Ε, προτείνω το εξής. Ένα 10% ως ε, πάγιο, αν θέλετε, άλλο ένα 10% να μοιραστεί μεταξύ των κομμάτων που συγκεντρώνουν πάνω από 1% στις ευρωεκλογέ και τα υπόλοιπα ανάλογα με την εκλογική δύναμη. Έκανα λοιπόν κάποιες προτάσεις, ο κύριος Βέμπερ ε, προχωρεί παραπέρα, όσον αφορά τώρα την ε, εξέταση αυτή. Κοιτάξτε, όσο εύκολα μπορεί να γίνει ένα κόμμα, ευρωπαϊκό κόμμα, εξίσου εύκολα θα πρέπει νομίζω και να συμβαίνει το αντίστροφο, γιατί βεβαίως στην αντίστροφη περίπτωση καταλήγουμε στα δικαστήρια κτλ. Επίσης τώρα για τα ζητήματα αξιών κτλ. Αυτά πρέπει να εξετάζονται εκ των προτέρων και με Κροάσεις κτλ. Γι' αυτό, κατά οποίο είναι σημαντικό κατά την ε, άποψή μου, θεωρώ πως ε, κάθε δραστηριότητα η οποία ε, έχει εθνικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα και θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να τι ακινδυνεύσει από την απαγόρευση κάποιου κόμματος δεν θα έπρεπε να σημαίνει. Δηλαδή εγώ θέλω πως δεν θα έπρεπε ε, να απαγορεύονται κόμματα. Γιατί, κοιτάξτε, και στις δημοτικές εκλογές ε, υπάρχουν κόμματα, μαζεύουν υπογραφές για να παραβούν το, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν, δεν το συζητάω αυτό. Και, τέλος, επειδή υπάρχει αυτό το μείγμα χρηματοδότησης 10, 15, 20 και 25% υπάρχει ε, ο μηχανισμός, κάποιος ο οποίος έλαβε χρήματα μα χρεωστήτως. να α, του αφαιρεθούν αυτά τα λεφτά το επόμενο έτος. Οπότε οτιδήποτε δίνεται πηγαίνει στην αντίστοιχη γραμμή του προπολισμού για το αντίστοιχο έτος και αναλόγως μετά εκεί επιστρέφεται κιόλας. Ε, Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Γεννάκου για να απαντήσει. Και η ποσότητα των τροπολογιών και οι ε, παρεμβάσει που ακούσαμε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικέ. Θα ε, κουράγιο, κυρία Γεννάκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που έγιναν. Θέλω όμως να θυμίσω κάτι δεν ανακαλύπτουμε σήμερα την πυρίτιδα. Σύστημα για τα ευρωπαϊκά κόμματα υπάρχει. Έστω και αν δεν υπάρχει στάτους. Δηλαδή η διαδικασία που περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αφορά στην αρμόδια επιτροπή, στην προκειμένη περίπτωση είναι η συνταγματικών υποθέσεων, η οποία μπορεί να κάνει ακροάσεις, να καλέσει τους ενδιαφερομένους από το κόμμα αυτό για το οποίο υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι δεν τηρεί τις αρχές και τα λοιπά. Ε, και η ενσυνεχεία διαδικασία είναι μέσα στα rules of procedure του Κοινοβουλίου, όπως έχουν σήμερα. Το Κοινοβούλιο προβλέπει στις, στον κανονισμό του και τα eminent persons, τα τρία πρόσωπα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την διαδικασία μέσω της αρμόδιας επιτροπής και τη διαδικασία μέσω της, ε, ε, της διάσκεψης των προέδρων και βεβαίως στο τέλος και αν χρειαστεί μπορεί το θέμα να πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο. Επομένως η θεωρία ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ελέγχει τα κόμματα κτλ. Κύριε Πρόεδρε δεν στέκει. Χρόνια τώρα το Κοινοβούλιο ελέγχει τα κόμματα. Δεύτερον, η εγγραφή των πολιτικών κομμάτων δεν πρόκειται να γίνεται σε πολιτικά πρόσωπα. Θα υπάρχει ένας αρμόδιος διοικητικός, ο οποίος θα εξετάζει τις προϋποθέσεις που αναφέρει το καθεστώς και εφόσον αυτές οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται θα κάνει την εγγραφή του κόμματος. Όμως το κοινοβούλιο ψηφίζει την αποδοχή των κομμάτων και αυτά δημοσιεύονται οι αποφάσεις αυτές στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτό γίνεται και σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Επομένως δεν πρόκειται να υπάρχει δίκη μηχανισμός όπου κάποιος θα ελέγχεται και κάποιος θα απορρίπτεται. Θα είναι μια διοικητική διαδικασία μέσα στο Κοινοβούλιο και θα γίνεται η εγγραφή. Αυτό που έχει σημασία είναι όταν υπάρξουν κατηγορίες και διαμαρτυρίες από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ότι ένα κόμμα δεν είναι δημοκρατικό τότε είναι διπλή η λειτουργία. Είναι οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, να κληθούν δηλαδή αυτοί να ακουστούν από την αρμόδια επιτροπή, να δώσει τη γνώμη της η αρμόδια επιτροπή και ταυτόχρονα μία ομάδα που έμειναν persons, τρία πρόσωπα λέει ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Νταφ λέει εννέα πρόσωπα να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε αυτό με την Επιτροπή. Επομένως υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, αν λάβετε υπόψη σας ότι εν τέλει υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε να έχουμε όλες τις διασφαλίσεις ότι ένα κόμμα δεν θα κριθεί με μεροληψία ή δεν θα κριθεί με ιδεολογικά κριτήρια. Διότι συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι δεν πρέπει ένα κόμμα να το δούμε ως αντίπαλο και να προσπαθήσουμε οι υπόλοιποι παραδείγματο χάρη να θεωρηθεί μη δημοκρατικό. Άλλωστε όλα αυτά είναι διαδικασίες που γίνονται φανερά κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι μυστικές διεργασίες και διαδικασίες. Δηλαδή η ανησυχία αυτή δεν έχει θέση εδώ. Σας επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά γίνονται χρόνια τώρα. Με κόμματα μάλιστα που δεν έχουν και απαραίτητο νομικό στάτους. Το δεύτερο ζήτημα που έθιξαν οι συνάδελφοι είναι το νομικό καθεστώς, αν θα είναι του κράτους μέλους ή όχι. Μα είναι σαφές κύριε Πρόεδρε. Αυτός ο κανονισμός δημιουργεί ένα στάτους ευρωπαϊκό. Μόνο ό,τι δεν ρυθμίζεται από αυτό τον κανονισμό μπορεί να ρυθμιστεί από την ομοθεσία του κράτους μέλους όπου το κόμμα έχει εγκατασταθεί. Επομένως ούτε διπλό καθεστώς υπάρχει, ούτε τέτοια. Υπάρχουν κόμματα με ευρωπαϊκό κανονισμό, όπως υπάρχουν συστήματα στα κράτη-μέλη που αποφασίζονται βάσει οδηγιών και κυρώνονται από τη Βουλή, πράγματα που δεν ρυθμίζονται από αυτόν τον κανονισμό θα ρυθμιστούν από το, την ομοθεσία των κρατών μελών όπου μπορεί να εγκατασταθεί το κόμμα. Και βεβαίως τα κόμματα πρέπει να έχουν την ελευθερία να εγκαθίστανται παντού. Αυτή η ελευθερία υπάρχει από τη συνθήκη του Μάστρακτ, κύριε Πρόεδρε. Ποιο μπορεί να εμποδίσει ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα να πάει όπου θέλει. Αυτό είναι προφανές, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως οι ανησυχίες για την εγγραφή, για το ρεζίστρ, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Το ρεζίστρ είναι διοικητική πράξη. Το κοινοβούλιο αποφασίζει όπως αποφασίζουν όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη κύριε Πρόεδρε, τα κόμματα εγγράφονται στο κοινοβούλιο. Ανεξαρτήτως της νομοθεσίας και από ποιο Υπουργείο προέρχεται κλπ. Τα κόμματα εγγράφονται στο Κοινοβούλιο. Και βεβαίως δεν είναι λογικό να ζητάμε η Επιτροπή ε, να έχει αυτή την αρμοδιότητα. Πού ακούστηκε η εκτελεστική εξουσία να έχει αρμοδιότητα για την εγγραφή των κομμάτων. Αυτό αν το πείτε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ε, θα σας πει ότι δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει διάκριση εξουσιών. Βεβαίω θα, υπάρχει, θα υπάρχουν από τα eminent persons ένας από την Επιτροπή, ένας από το Συμβούλιο, ένας από το Κοινοβούλιο ή και περισσότεροι όπως προτείνει ο κύριος Νταφ. Αυτό μένει να το εξετάσουμε αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν ανησυχίες. Ούτε έχει δημιουργηθεί τέτοιο θέμα ποτέ μέχρι σήμερα. Τώρα, ο διαχωρισμός των οικονομικών από την παρουσία των κομμάτων, όπως είπε ο κύριος Βίλαντ, βεβαίως υπάρχει είναι άλλο η αναγνώριση ενός κόμματος και άλλο η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση χωρίς εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Επομένως υπάρχει σαφέστατη διάκριση μεταξύ αυτών των δύο. Τώρα για τη μεταφορά κεφαλαίων που αναφέρατε κύριε Χέφνερ, αυτό ισχύει και για τα ιδρύματα. Ισχύει και για τα ιδρύματα για τη μεταφορά στο επόμενο έτος. Δεν ισχύει μόνο για τα κόμματα. Δείτε την έκθεση ε, καλά και θα το, θα το παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τώρα τα μέλη των κομμάτων. Ε, έγιναν διάφορες προτάσεις να είναι, λέει ο κύριος Ντάφ, να είναι ε, από 7 χώρες να είναι από 9 χώρες. Υπάρχουν άλλοι οποίοι λένε αντί να είναι από 7 χώρες να είναι από 4 χώρες. Τώρα το 7 χώρες κύριε Πρόεδρε είναι και στην πρωτοβουλία πολιτών έχει καθιδρυθεί και υπήρχε και στο προηγούμενο καθεστώς και εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο για το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Είναι, έχει διεθνή χαρακτήρα ένα κόμμα. Τώρα, εάν ένα ευρωπαϊκό κόμμα, κύριε Βίλαντ, μπορεί να κατεβεί σε όλες τις χώρες όπου έχει κόμματα μέλη, θα κατεβεί δια των κομμάτων μελών. Δεν μπορεί να κατεβεί ένα ευρωπαϊκό κόμμα ειδικό σε μια χώρα ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στις εκλογές. Και αυτό είναι και το λεπτό σημείο στο οποίο μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις με το Συμβούλιο. Ο σκοπός μας δεν είναι να υπονομεύσουμε την, ε, την παρουσία των ε, εθνικών πολιτικών κομμάτων. Απ' την άλλη πλευρά όμως δίνουμε τη δυνατότητα σε ε, μέλη των κοινοβουλίων ή των περιφερειακών κοινοβουλίων που δεν είναι μέλη κομμάτων, είναι ανεξάρτητοι βουλευτές ας πούμε να μπορούν και αυτοί να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Επομένως οι ανησυχίες που υπάρχουν νομίζω ότι δεν, δεν δικαιολογούνται. Πρώτον διότι όπως σας είπα και μέχρι σήμερα αυτή η πορεία ακολουθείται, δεν ανακαλύψαμε κάτι καινούριο και δεύτερον διότι τα πράγματα ισχυροποιούνται εφόσον θα υπάρχει ένα καθεστώς. Θα έρχεται λοιπόν στο κοινοβούλιο ο εκπρόσωπος του κόμματος και σε μια διοικητική αρχή, σε υπαλλήλους του κοινοβουλίου θα κάνει την εγγραφή του. Στο τέλος το κοινοβούλιο θα αποφασίζει ότι εγγράφονται όλα αυτά τα κόμματα εφόσον έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις. Η διοίκηση θα ξέρει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιο κόμμα πολιτικό, να θεωρηθεί ευρωπαϊκό. Δηλαδή διαδικασίες που ακολουθούνται πάντοτε και για όλα τα θέματα που αφορούν σε εμάς τους ίδιους. Και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι το Κοινοβούλιο θα έχει τόση μεροληψία και θα είναι τόσο υποκειμενικό ώστε θα θελήσει να εμποδίσει ένα κόμμα για να εγγραφεί ενώ το κόμμα αυτό θα είναι δημοκρατικό. Αυτά κύριοι συνάδελφοι είναι ε, κατά κάποιο τρόπο αυτοϋπονόμευση, δηλαδή προσβολή του εαυτού μας. Δεν μπορώ να τα δεχτώ εγώ ως εισηγήτρια ότι το κοινοβούλιο είναι μεροληπτικό. Είμαστε 754 βουλευτές από όλες τις χώρες, από εκατοντάδες κόμματα και δεν νομίζω πως αυτό ισχύει. Αντίθετα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιδείξει σε σχέση με όλες τις αρχές είτε αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε είναι Συμβούλιο, είτε είναι αρχές δημόσιες σε εθνικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγώ επιμένω ότι έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη ε, δημοκρατικότητα και ανοιχτή διαδικασία έχει επιδιώξει κάθε φορά την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και το βλέπετε και στα κράτη-μέλη. Επίσης βέβαια μέσα στον κανονισμό προβλέπεται και η συνεργασία με εθνικές αρχές. Δηλαδή δεν μπορεί να απαγορευτεί σε ένα κόμμα να εγγραφεί εάν δεν κληθεί το κόμμα αυτό να πει αν ισχύουν οι καταγγελίες που έχουν γίνει γι' αυτό ε, να γίνει ακρόαση ανάλογη, να υπάρξει η επιτροπή αυτή από τους σοφούς ε, και να εξεταστούν όλες οι διαδικασίες και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και να γίνει συνεργασία και με τις εθνικές αρχές. Επομένως δεν θα μείνει κανείς έξω από τη διαδικασία να έχει κάποιο λόγο επί του θέματος. Δεν είναι μόνο το Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι αυτό είναι, είναι προφανές, δηλαδή τα κόμματα εγγράφονται ε, στο κοινοβούλιο και δεν υπάρχει θέμα να είναι ιδεολογικού χαρακτήρα όλα αυτά. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω και τη σοσιαλιστική ομάδα διότι πράγματι 14 τροπολογίες που έχουν γίνει είναι τροπολογίες για τις οποίες μπορούμε να συνεννοηθούμε αλλά και άλλους συναδέλφους και νομίζω ότι αν ε, εξαλείψουμε τους φόβους μας για την εγγραφή του κόμματος και για το ποιος θα ελέγχει και συνεννοηθούμε για τα οικονομικά, εγώ επιμένω στο 10-90, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι 90% πρέπει να είναι βάση ε, των ποσοστών και το 10% να διανέμεται εξίσου ε, τότε βεβαίως μπορεί να είναι 370 οι τροπολογίες αλλά δεν θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σύντομα ένα κείμενο το οποίο θα διαπραγματευτούμε με αποτελεσματικότητα και επιτυχία στο, ε, με το Συμβούλιο και την ε, Επιτροπή. Και βεβαίως ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους διότι από την άλλη πλευρά οι πολλές τροπολογίες δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι το αναμένουν και στα κράτη-μέλη με ενδιαφέρον και κυρίως οι πολίτες που όπως είπαμε κύριοι συνάδελφοι αυτό δεν θα υπολογίζεται στη χρηματοδότηση. Τα μέλη που εγγράφονται στα ευρωπαϊκά κόμματα θα τα υπολογίζουν τα ίδια τα κόμματα στα συνεδριά τους και στον τρόπο λειτουργίας τους. Όμως δεν θα υπολογίζονται στη χρηματοδότηση γιατί τότε βέβαια τα κόμματα θα έτρεχαν να γράψουν εκατομμύρια πολίτες για να μπορέσουν να πάρουν περισσότερη χρηματοδότηση. Άρα και εδώ υπάρχει μία ρήτρα η οποία αποκαθιστά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γεννάκου. Θα ψηφίσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 19 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα όμως να μας πείτε αν θεωρείτε ότι πρέπει να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία στις 19 Φεβρουαρίου ή αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει μία ακόμα συνάντηση με την ελπίδα να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική τροπολογία για να μας διευκολύνει και λίγο τη ζωή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε μία ημερομηνία για μία έκτακτη συνεδρίαση στη διάρκεια της συνεδρίασης του, ε, το Φεβρουάριο. Θα ήθελα να ακούσω την απόψή σα. Θα κάνουμε μια ενδιάμεση συνεδρία. Οπωσδήποτε κύριε Πρόεδρε, ε, θα πρέπει να γίνει. Μπορούμε τη Δευτέρα να την κάνουμε αυτή στο Στρασβούργο. Οπωσδήποτε πρέπει να ξαναβρεθούμε όλοι να συζητήσουμε. Και εντωμεταξύ θα έχω και εγώ επιχειρήσει, θα δω και τους shadow rapporteurs, ε, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε συμβιβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε όλοι. Νομίζω ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι. Επομένως, αυτό θα κάνουμε. Θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο ζήτημα τη Δευτέρα του Στρασβούργου, δηλαδή στις 4 Φεβρουαρίου. Και η ψηφοφορία παραμένει για τις 19 Φεβρουαρίου. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη έχουμε το θέμα της τροποποίησης του κανονισμού 35483 για τα ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την, ε, ε, ε στο Πανεπιστήμιο της ε, Φλωρεντίας, αλλά επειδή είναι ήδη πάρα από τις 5, προτείνω να ψηφίσουμε πρώτα και για όσους ήρθαν λίγο καθυστερημένα υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε μόνο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών γιατί οι ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές αποφασίσαμε να αναβληθούν για αύριο το πρωί στις 10 υπό την επιφύλαξη διαφορετικής άποψης από τη συνεδρίαση των συντονιστών η οποία δεν θα γίνει σήμερα αλλά θα γίνει αύριο το πρωί από τις 9 μέχρι τις 10. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης για το 2013. Αν είστε έτοιμοι, τροπολογία 1 του κυρίου Νταφ για την παράγραφο 6. Υπέρ. Θέλετε το λόγο κύριε Νταφ ή θέλετε να ψηφίσουμε μόνο. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Να μετρήσουμε γιατί δεν βλέπω όλο το κόσμο τα χέρια του. Ποιος είναι υπέρ τη τροπολογία 1 του κυρίου Νταφ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 2 για την παράγραφο 7 και πάλι του κυρίου Νταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μία αποχή. Τροπολογία 3 στην παράγραφο 16 αυτή αποσύρθηκε. Αποσύρεται, έτσι δεν είναι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 4 στην παράγραφο 17 και πάλι από τον κύριο Ντάφη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα το σύνολο του εγγράφου. Υπέρ για τελική ψηφοφορία. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Κατά. Κανείς δεν είναι κατά. Αποχές. Μία αποχή. Δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν με 12 ψήφους υπέρ, καμία κατά και δύο εποχές. Καλώς. Ευχαριστώ τον κύριο Ραντζέλ. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Τροποποίηση του κανονισμού 354-83 σχετικά με την κατάθεση των ιστορικών αρχείων των θεσμικών οργάνων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Όπως γνωρίζετε, Η νομική βάση για την υπόθεση αυτή είναι στο άρθρο 352 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε δεν είναι η τροποποίηση ή η κατάθεση τροπολογιών, απλώς εκφράζουμε κατά πόσον εγκρίνουμε την πρόταση του Συμβουλίου. Αρχικώς μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού είχαμε σκοπό να παρέμβουμε με μια ενδιάμεση έκθεση για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και την άποψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά από κάποιες άτυπες συναντήσεις ε, μας συμβουλεύτηκε να συστήθηκε να μην κάνουμε διάμεση έκθεση, αλλά να παρουσιάσουμε απλώ τη γνώμη μα όταν θα είναι έτοιμο το έγγραφο του Συμβουλίου. Τι ανησυχίε που έχουμε και εμεί εδώ, και εγώ συντάκτη τη γνωμοδότηση, αλλά και η πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτισμού, είναι κατά πόσον μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι από νομική ε, και οικονομική σκοπιά ε, η κατάθεση των ιστορικών αρχείων στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της θα μπορούσε να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Από ό,τι φαίνεται μας δίνονται αυτές οι εγγυήσεις. Υπήρχε και η ελπίδα να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για την κατανομή των δαπανών για τα διάφορα θεσμικά όργανα που καταθέτουν τα ιστορικά τους αρχεία ε, στην, ε, στο Ινστιτούτο. Από ό,τι φαίνεται και ε, προς τα εκεί προχωρούμε με αρκετή σαφήνεια. Η Ιταλία διαθέτει τους χώρους, αλλά από εκεί και πέρα τα θέματα της διαχείρισης και την κατάθεση των αρχείων προϋποθέτει και την οικονομική συνδρομή και άλλων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια και να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση και ελπίζουμε να υπάρχει είναι εύκολη η χρήση των αρχείων, επομένως να μην υπάρχει μόνο κατάθεση εγγράφων, αλλά να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονική κατάθεση, είτε να υπάρχουν αντίγραφα ή κάτι αντίστοιχο. Είμαστε εν αναμονή του εγγράφου όμως του ε, Συμβουλίου. Από ό,τι φαίνεται όλα βαίνουν καλώς. Εμείς λοιπόν προς το παρόν θα ετοιμάσουμε μια πολύ σύντομη έκθεση, η οποία απλώ θα εκφράζει την έγκριση ή την απόρριψη του εγγράφου του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω αν κάποιο θέλει το λόγο. Αν ναι, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν βλέπω κάποιον να θέλει να παρέμβει. Αναμένουμε λοιπόν το έγγραφο του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 35483 για την κατάθεση των ιστορικών αρχείων των θεσμικών οργάνων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερησία διάταξη. Ωραία λοιπόν. Όπως είπαμε επανειλημμένως, αναβάλλεται η συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα λόγω της υποχρεωτικής απουσίας είτε λόγω πτήσεων είτε λόγω άλλων υποχρεώσεων των κυρίων Τρασκόφσκι και Γκουαλτιέρη και θα γίνει αύριο το πρωί στις 9 συνεδρίαση των συντονιστών και η συνεδρίαση ε, η τακτική θα ξεκινήσει στις 10. Από τις 10 έως τις 12 ε, και 11 συγγνώμη, θα συνεδριάσουμε γιατί στις 11 θα έρθει η Ιρλανδή Υπουργός. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Πέρασε τη συνεδρία σας.